Uh, Καλησπέρα σας. Ας ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Η πρόεδρος μας, η κυρία Μπόλς, μου ζήτησε να λάβω την προεδρία της συνεδρίας αυτής για την πρώτη έκθεση και θα ακούσουμε στη συνέχεια Μάλλον στη συνέχεια θα με διαδεχθεί ο κύριος Κυκλούνα αφού παρουσιάσει την έκθεσή του. Σας ζητώ συγγνώμη για την αλλαγή αυτή στο πρόγραμμα. Πρέπει πάντως να συνεχίσουμε τις εργασίες μας στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Ας ξεκινήσουμε με την έκθεση για την οποία είμαι εγώ εισηγητής, αναφέρομαι στο πρόγραμμα Φισκάλης 2014-2020 και προβλέπεται μία ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τις τροπολογίες. ...54 συνολικά είναι τροπολογίες. Τροπολογίες τις οποίες διάβασα... ...και μπορώ να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα... γιατί πολλές από τις τροπολογίες αυτές που κατέβαλαν οι συνάδελφοι επικεντρώνονται στο πολύ βασικό ζήτημα της ενίσχυσης της μάχης κατά της φοροδιαφυγής, της φορολογικής απάτης. Οι τροπολογίες επικεντρώνονται λοιπόν στην καταπολέμηση αυτών των πολύ αρνητικών συμπεριφορών. Συμφωνώ λοιπόν με όλες αυτές τις τροπολογίες οι οποίες επικεντρώνονται σε αυτά τα ζητήματα, φορολογική απάτη, φοροδιαφυγή και χαίρομαι ιδιαίτερα που οι συνάδελφοί μου συμφώνησαν να υπογραμμίσουμε τα στοιχεία αυτά στην έκθεσή μου. Θα συνεργαστώ με τους πιο δυσηγητές και με τους άλλους συναδέλφους τις επόμενες εβδομάδες προκειμένου να καταλήξουμε και σε συμβαστικές τροπολογίες. Βλέποντας την έκθεσή μου και τις προτινόμενες τροπολογίες, πιστεύω ότι πραγματικά μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν πολύ καλό συμβιβασμό. Υπάρχουν βέβαια και άλλες τροπολογίες, τις οποίες θα πρέπει να τις εκτετάσουμε περισσότερο και τις οποίες θα πρέπει να ομαδοποιήσουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Αναφέρομαι σε τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που παρακολουθούμε την εφαρμογή του προγράμματος αυτού πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε την υλοποίηση του προγράμματος κατά την εφαρμογή του. Αυτό απασχολεί συγκεκριμένες τροπολογίες και πιστεύω ότι αυτές θα πρέπει να ομαδοποιηθούν σε συμβαστικές τροπολογίες. Ωστόσο υπάρχουν και ορισμένες τροπολογίες τις οποίες πρέπει προσωπικά να συζητήσω με τους συναδέλφους που τις υπέβαλαν Νομίζω ότι ορισμένε από τι τροπολογίε αυτέ είναι θετικέ, μπορούμε να τι υποστηρίξουμε, απλώ θα πρέπει να δούμε αν τελικά οι τροπολογίε αυτέ πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το κείμενο ή σε κάποιο άλλο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, σε τι τροπολογίες αναφέρομαι. Ο σταδελφός μας, ο κύριος Φιλίπ Λαμπέρ, πρότεινε στην τροπολογία υπαριθμών 21 Κράτη-μέλη τα οποία προχωρούν σε διασυνοριακές φορολογικές συναλλαγές να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα πρέπει η τροπολογία αυτή να ενταχθεί σε αυτή την έκθεση. Εφόσον η έκθεση αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα στην εφαρμογή ενός συγκεκριμένου προγράμματος. Ενδεχομένως η τροπολογία σας να μπορούσε να συμπεριληφθεί σε μια άλλη έκθεση, σε μια έκθεση που θα είχε να κάνει με την συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η συγκεκριμένη έκθεση δεν έχει να κάνει με την ενίσχυση της υποχρέωσης των κρατών μελών να υποβάλουν εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως μπορούμε και αυτό να το συζητήσουμε. Υφίστανται λοιπόν ορισμένες τροπολογίες, τις οποίες πιστεύω ότι θα πρέπει να αναλύσουμε λίγο περισσότερο, να συζητήσουμε περαιτέρω με τους κοιόδης συγητές και με τους βουλευτές που τις πρότειναν προφανώς. και νομίζω ότι δεν θα πρέπει στην συγκεκριμένη έκθεση που εξετάζουμε να προσπαθήσουμε να εντάξουμε συστάσεις ή άλλες σχετικές τροπολογίες οι οποίες ε, σχετίζονται με συγκεκριμένους κανονισμούς. Υπάρχει μία ακόμα τροπολογία, αυτή του κυρίου Βολφ Κλίνγκ, η τροπολογία 63, τροπολογία που έχει να κάνει με το ποσό των χρημάτων που δίνεται στο πρόγραμμα αυτό. Ξέρετε ότι στο πρώτο τμήμα της έκθεσης λέγεται ότι το ποσό για το πρόγραμμα αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης. Λέμε ότι το ποσό χρηματοδότησης θα οριστικοποιηθεί μετά το τέλος των πραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και επομένως το ποσό αυτό για το πρόγραμμα φυσκαλής θα εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις, από την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο κύριος Κλίνς ανταυτού στην τροπολογία 63 μας προτείνει να λάβουμε υπόψη μας την συμβολή των κρατών μελών Πρέπει να το συζητήσω περαιτέρω αυτό μαζί του για να καταλάβω τελικά τι είχε κατά νου όταν κατέθεσε αυτή την τροπολογία. Πέρα από αυτά νομίζω ότι ε, μπορούμε να επεξεργαστούμε τις υπόλοιπες τροπολογίες και να καταλήξουμε τελικά σε ξεκάθαρες συμβαστικές προτάσεις για την Επιτροπή μας. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό και θα ήθελα να ακούσω τώρα την άποψη των σκιωδών εισηγητών και ξεκινώ με τον κύριο Χουάνκ Νόγκ, ο οποίος εκπροσωπεί τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ε, πράγματι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Ως προς αυτό το σχέδιο έκθεσης πρέπει να πω ότι δεν είναι δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναπροσδιορίσει πλήρως το φισκάλις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή η οποία έχει τις ε, ικανότητες να το κάνει αυτό. Εν εμείς έχουμε την ευθύνη να θεσπίσουμε ασφαλιστικές δικλίδες, ώστε τα κονδύλια που θα έχει το πρόγραμμα να δαπανώνται με τον πιο δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. Και αυτό ισχύει κυρίως ως προς τη συμμετοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς τις μη επιλέξιμες δράσεις, ως προς το συντελεστή συγχρηματοδότησης, ως προς την ε, ε, έκκληση σε εξωτερικούς ε, αξιολογητές και εμπειρογνώμονες και ως προς τον έλεγχο εκ των υστέρων του προγράμματος. Συμφωνούμε με τον εισηγητή και τον σκιώδη εισηγητή. Οι υποψήφιες χώρες που, και οι χώρες που είναι σε φάση προσχώρησης θα πρέπει να μπορούν να συμμετάσχουν χωρίς περιορισμούς. Όμως, όταν εντάσσονται στην πολιτική γειτονία θα πρέπει να συμμετέχουν μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή. Ως προς τις ε, ε, δράσεις ε, τις μη επιλέξιμες πιστεύω ότι πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένες παράγραφοι. Η παράγραφος 9 του άρθρου 7 πιο συγκεκριμένα γιατί έτσι όπως είναι διατυπωμένη αυτή τη στιγμή επιτρέπει τη χρηματοδότηση οποιοδήποτε σχεδόν πράγματος και αυτή την έννοια έχει και η τροπολογία υπαριθμών 58 που υποβάλλω. Μέχρι το 100% είναι ο συντελιστή συγχρηματοδότησης από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να περιοριστεί στο 80%. Κάτι το οποίο είναι λογικό για να συνάδει και με αυτό που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα άλλα προγράμματα που έχουν να κάνουν με το Ταμείο Συνοχής και βέβαια να κρατηθεί το 100% για τις χώρες που λαμβάνουν οικονομική βοήθεια. Ως προς τις εξωτερικές δράσεις, καλό θα ήταν να έχουμε τα κράτη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να μην διευρύνουμε εκεί την εκπροσώπηση και ε, με εκπροσώπους τρίτων χωρών. Τροπολογία 37, 38, 39, 40. Αυτές οι τροπολογίες αφορούν σε αυτό το θέμα. 45, 48, 67 και 68, οι τροπολογίες μου αυτές θέλουν να θεσπίσουν ξεκάθαρες αρχές για την αξιολόγηση και την εξέλιξη του προγράμματος, το οποίο πρέπει να αξιολογείται βάσει αριθμημένων δικτών, βάσει αποτελεσμάτων της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής. Να μην βασίζεται η αξιολόγηση μόνο στις μαρτυρίες των συμμετεχόντων και ε, θα πρέπει να τεκμηριώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα αυτά. Έχουμε σύγκληση και με τις άλλες πολιτικές ομάδες πάνω σε πάρα πολλά θέματα, πολλές τροπολογίες και είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε σε μια πολύ καλή συμβιβαστική λύση ως προς το σχέδιο κανονισμού αυτό. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βολφ Λίντς, αλλά πρώτα ε, αλλά είναι ο κύριος Σμίτ εδώ και θα μιλήσει εξ ονόματός του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε εισηγητά. Ναι, εγώ τώρα είμαι ο κύριος Κλίνς για τώρα. Ε, δια του στόματός μου λοιπόν ο κύριος Κλίνς θέλει να σας ευχαριστήσει για τη δουλειά που κάνετε, θέλει να εκφράσει την εμπιστοσύνη του. Ε, πιστεύει ακραδάντως ότι το αποτέλεσμα θα βοηθήσει όλους μας και θα είναι πολύ καλό. έχει υποβάλει κάποιες προτάσεις τροποποίησης του κειμένου και επειδή καθυστέρησα λόγω των αλλαγών προγραμμάτων δεν μπόρεσα να ε, ακούσω αν ήδη έχετε σχολιάσει αυτές τις προτάσεις αλλά θα το κάνω ούτως ή άλλως. Εξωτερικοί εμπειρογνώμονες πρέπει να εμπλακούν όπου δει για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος φυσκάλης και να μην αποκλειστούν πλήρως όπως προτείνεται από τον εισηγητή. Αυτό Αυτά λοιπόν και βλέπω ότι σε αυτό το σημείο διαφωνείτε με τον κύριο Κλάιντς. Η κατανομή πόρων στο πρόγραμμα συγκεκριμένη δράση, εξοπλισμό τεχνολογία πληροφορική θα πρέπει να γίνονται με ισόρροπο, ισορροπημένο τρόπο και να μην περιορίζεται με τον τρόπο που υποδεικνύει ο εισηγητή. Δεύτερο σημείο διαφωνία κύριο Κλίντ και ημών Ε. ε. Ω προ την εφαρμογή του προγράμματο φυσκάλης, το, ο φόρτος, ο οικονομικός θα καθοριστεί ανάλογα με τη συνεισφορά και τη συμβολή του κάθε κράτος μέλος. Και θα πρέπει να υπάρχουν εκθέσεις αξιολόγησης οι οποίες θα πρέπει να καταρτίζονται τουλάχιστον άπαξ ετησίως. Αυτά προς το παρόν σας ευχαριστώ και είμαι σίγουρος και ελπίζω ότι θα φτάσετε σε συμβαστική λύση εσείς ως εισηγητής ε, σε συνεργασία με τον κύριο Κλίντς. Ευχαριστώ ο κύριος Φιλίπ Λάμπερτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, εγώ παίζω όλους τους ρόλους σήμερα. Ε, ελπίζω αύριο να απαλλαγώ. Φτάνει μία μέρα. Γιατί, ε, εν πάση περιπτώσει, μέχρι αύριο θα έχει γεννήσει η σύζυγος ε, του κυρίου που θα αντικαταστήσω που αντικαθιστώ τώρα με την παρέμβασή μου. Ε, να πω λοιπόν ότι είμαστε εδώ σε μια κάπως ειδική κατάσταση. Πώς ερμηνεύεται η απουσία τόσων συναδέλφων εδώ, μόνο ως ένδειξη εμπιστοσύνης στα δικά μας πρόσωπα εμείς που διαχειριζόμαστε αυτό το πολύ δύσκολο φάκελο. Όταν έχουμε λοιπόν μια τόσο ανοιχτή δημόσια επίδειξη εμπιστοσύνης και πίστη στο πρόσωπό μας πρέπει να την υπογράψουμε. Ε, σας καλώ λοιπόν όλους για λίγα δευτερόλεπτα να βιώσουμε αυτή την απόλαυση για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μας αφού λείπουν όλοι αυτοί εδώ σήμερα από αυτή την αίθουσα. Από εκεί, κύριε, πέρα κύριε Πρόεδρε, το φυσκάλις δεν μπορεί να κάνει τα πάντα και να πετύχει τα πάντα. Είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών και το θέμα είναι πώς θα το ενθαρρύνουμε, πώς θα ενθαρρύνουμε αυτή τη συνεργασία. Πρέπει να τονίσω την ανάγκη όχι μόνο για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τους φορολόγουμένους, αλλά και ανταλλαγή πληροφοριών για τις φορολογικές διατάξεις και αποφάσεις και αυτό είναι το βασικό για να προλάβουμε τη φοροδιαφυγή από μεγάλες επιχειρήσεις. Η περιβόητη λέξη που αρχίζει από C, conditionality, από α δηλαδή στα ελληνικά, αιρεσιμότητα, είναι η λέξη καραμέλα στο στόμα των Γερμανών και του κυρίου Ντράγκη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εάν θέλεις ε, να ε, ενταχθείς θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένου όρους και προϋποθέσεις. Βεβαίω οφείλουμε να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών και για φορολογουμένους και για τις αποφάσεις τις φορολογικές. Τώρα, ως προς τους εμπειρογνώμονες. Ναι. Εάν καλέσουμε εμπειρογνώμονες, δεν θα ήθελα, θα είχα πολλές επιφυλάξεις ε, να επιλέξουμε εμπειρογνώμονες μόνο από τον επιχειρητικό, επιχειρηματικό κόσμο. Σίγουρα την ξέρουν τη δουλειά, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι έχουν και τους ίδιους στόχους με μας μόνο. Καλό θα ήταν να έχουμε επιρογνώμονες, πολύ καλά καταρτισμένους, αλλά και από άλλους κύκλους, από άλλες κοινότητες, όχι μόνο από την επιχειρηματική κοινότητα. Ε, εκπροσώπους της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών που έχουν πράγματι εμπειρογνωμοσύνη στα τομέα της φορολογίας. Και σίγουρα η ικανότητα καταπολέμησης φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής είναι αυτό που πρέπει να οικοδομήσουμε. Είναι και δύσκολο να επιτευχθεί. Στόχος που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ο εξής. Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο για να αυξήσουμε και το μέγεθος και την αποτελεσματικότητα ποιότητα των δημοσίων λειτουργούν που πραγματικά βγάζουν τη δουλειά, που πραγματικά καταπολεμούν τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη. Αυτές είναι οι βασικές μου παρατηρήσεις. Δύσκολο θα είναι, θα χρειαστεί ίσως, θα χρειαστούμε 10 ή 12 συνεδριάσεις με τους κοιόδες εισηγητές και τον εισηγητή, αλλά πιστεύω ότι τελικά θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ίσως 12 να μην μπορέσω ο ε, Κύριε Σιγητά, αν συμφωνήσετε με όλες μα τι τροπολογίες, δεν χρειάζεται καν να συναντηθούμε ούτε μία φορά, πόσο, ή μάλλον 12. Ο πρόεδρο, ευχαριστώ κύριο Στρίετ. Καλησπέρα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην αρχή της απογευματινής μας συνεδρίασης σκέφτηκα το εξής. Μια ωραία ήρεμη απογευματινή συνεδρίαση ε, ευκαιρία για καφέ, αλλά ο Φίλιπ το έθεσε πολύ κέρια το ζήτημα με αυτά που μας είπε και συνειδητοποίησε ότι έχει δίκιο είναι η συνεδρίαση μεταξύ ημών. Εμείς έχουμε τη μεγαλύτερη επιρροή, σε εμά έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη όλοι, είμαστε οι περισσότερο αξιόπιστοι, όλα τα μέλη της Επιτροπής Οίκων εμπιστεύονται εμάς και τα πρόσωπά μας, γι' αυτό και λείπουν. Άρα μπορούμε πράγματι να αποφασίσουμε ό,τι θέλουμε και αυτοί θα ακολουθήσουν. Δηλαδή τι εννοείται λέει ο Φίλιππ, ότι είναι ετεμπέληδες ή ενδεχομένως μειωμένων νοητικών προσόντων ε, απαντάει ο μιλητή. Μπορούμε να το συζητήσουμε σε άλλο, ε, κάποια άλλη στιγμή. Έχουμε πολύ χρόνο, μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Θα ήθελα να κάνω 5-6 ε, γενικές ε, παρατηρήσεις. Όπως γνωρίζετε, εμείς είμαστε κάπως επιφυλακτικοί με προγράμματα τύπου φισκάλης. Με χαρά όμως διαπιστώνω και ομολογώ ότι η πλειονότητα των προσεγγίσεων και των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί είναι αρκετά κοντά στη δική μας νοτροπία. Αυτό καταρχάς. Ε, να πω ότι συμφωνούμε απολύτως με την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής. Εγώ έχω υποβάλει τροπολογίες για καλύτερη διατύπωση του κειμένου, δεν είναι καθόλου σημείο διαφωνιών αυτό και υπ' αυτή την έννοια Έρχομαι στο σημείο 2 της παρέμβασής μου. Διασυνοριακές απάτες. Εμείς πιστεύουμε ή θα θέλαμε να πιστεύουμε, εν πάση περιπτώσει, ότι προγράμματα τύπου φυσκάλης πράγματι βοηθούν στον περιορισμό της διασυνοριακής απάτης. Ένα φαινόμενο το οποίο πλήττει τον ανταγωνισμό και την ανάπτυξη και το οποίο μπορεί μάλιστα να περιορίσει και την ανάπτυξη. Τρίτη παρατήρησή μου είναι η εξή: Κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού των φορολογικών διοικήσεων. Έχω υποβάλει νομίζω δύο ή τρεις τροπολογίες που ε, τονίζουν αυτή την ανάγκη. Και το λέω αυτό διότι η εθνική η φορολογική διοίκηση διαφέρει από χώρο σε χώρα. Για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τη φορολογική απάτη θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε καλύτερα τους ανθρώπους, να έχουν περισσότερες γνώσεις η ε, λειτουργεί της φορολογικής διοίκησης στα διάφορα κράτη-μέλη. Και θυμάμαι και τη σύντηση με τον κύριο Κλίντς. Ε, κινούμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ο κίνδυνος υπερβολικής σπατάλης χρημάτων. Και αυτό δεν ε, ε, έρχεται σε, καθο... σε καμία αντίθεση με αυτό που έχουν πει άλλοι. Έκτον, εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. Καταλαβαίνω ότι Ε, μπορεί να υπάρχει θέμα, αλλά εμείς είμαστε υπέρ των εξωτερικών υπορογνωμών υπό τον όρο ότι ο κατάλογος είναι δημόσιος, ότι υπάρχει διαφάνεια, ότι γίνεται ενημέρωση σε τακτά χρονικά διαστήματα του καταλόγου, αλλά και της διαδικασίας βάσει της οποίας, της οποίας επιλέγονται αυτοί οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια εκεί και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι καλοί εμπειρογνώμονες βεβαίως και στοιχίζουν. Αυτές είναι οι βασικές μου παρατηρήσεις και τέλος θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά το γεγονός ότι είμαστε σχεδόν στο ίδιο μήκος κύματος ε, σε γενικές γραμμές. Επομένως δεν φαντάζομαι να υπάρξουν δυσκολίες ε, για την επίτευξη τελικού συμβιβασμού. Ευχαριστώ. Έχουμε και άλλων ένα τον κύριο Χουντή, τον κύριο Νικόλα Χουντή, αλλά δεν είναι παρόν. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να μιλήσει εξ ονοματός του. Από ό,τι φαίνεται όχι. Άλλοι συνάδελφοι, επιθυμεί κάποιος άλλος ενδεχομένως να λάβει το λόγο. Πολύ ωραία. Τότε επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΚΟΝ είναι προγραμματισμένη για τις 28-29 Νοεμβρίου και στην Ολομέλεια ε, προβλέπεται να ψηφίσουμε το Μάρτιο του επόμενου έτους ε, ανάλογα με την έκφαση που θα έχει η τριμερή συζήτηση. Δεν θα πάμε στην Ολομέλεια πριν έχουμε ολοκληρώσει την τριμερή συζήτηση με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Πω, πω. Δυστυχώς πρέπει να διακόψουμε μέχρι τις 4 και 20 μέχρι να έρθει ο κύριος Σικλούνα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω απλά να αναφέρω ότι επειδή εγώ θα ξανάρθω στις 4 και 20, κοιτάξτε, είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι εδώ από το άλλο κτίριο μέχρι εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω <laughs> το Προεδρείο για την ευκαιρία που μας δίνει να γυμναστούμε λιγάκι, καθότι η δουλειά μας είναι καθιστική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη για τις αλλαγές στο πρόγραμμα. 4 και 20 λοιπόν. Αν έχει την καλοσύνη να είστε και πάλι εδώ. Έτσι θα Yes, we can start. I will be chairing this uh, point four, which uh, concerns. Uh, Καλησπέρα σας. Θα προεδρεύσω εγώ για το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, σχέδιο έκθεσης για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Πρόκειται για την τροποποίηση του κανονισμού 223 κάθετος 2009. Σας ζητώ συγγνώμη που έφτασα καθυστερημένος. Έφυγα από το σπίτι στις 6.30 το πρωί και υπήρχαν πολλές καθυστερήσεις όμως με τις πτήσεις. Γι' αυτό το λόγο έφτασα τόσο καθυστερημένος. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε πάντως. Να σας περιγράψω καταρχάς αυτό το σχέδιο έκθεσης το οποίο παρουσίασα. Και να σας πω κάτι ακόμα. Αφού ολοκληρώθηκε αυτό το σχέδιο έκθεσης και κοιτώντα το με κάποια απόσταση, μπορώ να σας πω ότι είμαι κάπως απογοητευμένος με τον εαυτό μου. Γιατί το λέω αυτό, θεωρώ ότι δεν προχώρησα αρκετά. Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία που μας δίνεται για να μιλήσουμε για την βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών δεδομένων. Ξέρετε ότι πολύ συχνά κατά τρόπο ανεπίσημο λέμε ότι τα στατιστικά δεδομένα θα πρέπει να έρχονται εγκαίρως, θα πρέπει να είναι συγκρίσιμα και ακριβή και θεωρώ ότι όντως θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσει αυτές γιατί σίγουρα τα στατιστικά δεδομένα αποτελούν πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς. Πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, για πολλά ενδιαφερόμενα μέρη εν γέννη. Ωστόσο, πολύ συχνά μιλάμε για την ε, έκβαση τελικά, για το τελικό αποτέλεσμα. Όταν έχουμε τα στατικά δεδομένα στα χέρια μας, έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να βελτιώσουμε την όλη διαδικασία κατάρτισης και διάχυσης αυτών των ευρωπαϊκών στατιστικών δεδομένων. Αυτός είναι ο στόχος αυτής της ε, έκθεσης. Τα τελευταία χρόνια το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα έχει πλέον μια καλύτερη διακυβέρνηση και επομένως το όλο σύστημα εφαρμόζει τα απαραίτητα κριτήρια αποτελεσματικότητας και ποιότητας. Υπάρχει ένας διοντολογικός κώδικας και προβλέπονται επίσης πάρα πολλά μέσα ελέγχου. Και εν γέννη όλα αυτά τα κριτήρια έχουν βοηθήσει όλες τις χώρες οι οποίες εμπλέκονται στο ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε ορισμένα παραδείγματα όπως αυτό της Ελλάδας. Εξετάζοντας την περίπτωση της Ελλάδας βλέπουμε ότι τα όσα έχουν γίνει δεν ήταν αρκετά. Υπήρξε μία συστημική αποτυχία, μπορούμε να πούμε, μια αποτυχία στα πλαίσια του συστήματος αυτού. Καλούμεθα λοιπόν να αναλάβουμε δράση προκειμένου να διορθώσουμε τις αδυναμίες του συστήματος, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν νέους συστημικούς κινδύνους. Γι' αυτό λοιπόν μας, ζητάτε, μας ζητείτε να αναλάβουμε δράση. Μετά την ε, ελληνική οικονομική κρίση, σε πολλές χώρες παρατηρείται πλέον πάρα πολύ αυστηρά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει το σύστημα αυτό να βελτιωθεί και ότι θα πρέπει οι επιμέρους εθνικές στατιστικές υπηρεσίες να είναι όλο και πιο αυτόνομες και ανεξάρτητες. Μας ζητήθηκε επίσης να μην αντιδρούμε μόνο εκ των υστέρων, αλλά μας σε θέση να αντιμετωπίσουμε εκ των προτέρων κάποια προβλεπόμενα προβλήματα. Το εφιστάμενο σύστημα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ανανεωθεί γιατί ουσιαστικά είναι παγιωμένο μέσα στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Μόνο αν τροποποιηθεί η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν ουσιαστικά να δυναμωθούν τα στοιχεία ποιότητας του υφιστάμενου συστήματος του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, προκειμένου αυτό να γίνει τελικά πιο ανεξάρτητο. Πιστεύω ωστόσο ότι υπάρχει ακόμα ένα περιθώριο στα πλαίσια του φυστάμενου συστήματος να επιφέρουμε κάποιες αλλαγές. Μπορεί κάποιες αλλαγές να είναι αυτορυθμιζόμενες. Στο κείμενο λοιπόν αυτό προσπαθούμε να δούμε αν μπορούμε τελικά να πείσουμε τους χρήστες των στατιστικών αυτοδεδομένων... ότι μετά τη δική μας την επέμβαση θα είναι αδύνατον πλέον να δούμε παραδείγματα σαν το ελληνικό. Αυτό είναι το διακύβευμα Κατά αυτόν τον τρόπο πρόκειται να μας αξιολογήσουν. Το νομικό καθεστώς του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος είναι σαφώς πιο αδύναμο αν το συγκρίνουμε με το ευρωπαϊκό σύστημα το οποίο ισχύει για τις κεντρικές τράπεζες, για παράδειγμα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να συγκρίνουμε το σύστημα αυτό με ανάλογα ευρωπαϊκά συστήματα για τα οποία έχουμε μια κάποια εμπιστοσύνη. Ξέρω ότι ε, πολύ συχνά οι συγκρίσεις οδηγούν σε κάποια λανθασμένα συμπεράσματα, αλλά και πάλι δεν μπορούμε να πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα αυτή τη στιγμή βρίσκεται πραγματικά στο ποιοτικό επίπεδο το οποίο έχουμε για το σύστημα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αν συγκρίνουμε, για παράδειγμα, τα όσα ισχύουν για τη Eurostat και όσα ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το ίδιο και για τα εθνικά στατιστικά όργανα που είναι ουσιαστικά υπηρεσίες κυβερνητικές που υπάγονται τελικά σε συγκεκριμένα υπουργεία και έχουν προπολογισμό τον οποίο αποφασίζουν εθνικά κοινοβούλια και εθνικές κυβερνήσεις. Η εθνική κυβέρνηση λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένε γραμμές του προπολογισμού προκειμένου να ελέγξει και να επηρεάσει τη στατιστική της υπηρεσία. Πρέπει λοιπόν οι ε, εθνικές στατιστικές υπηρεσίες να γίνουν όλο και πιο αυτόνομες, ανεξάρτητες υπηρεσίες και ουσιαστικά να παράγουν ένα εθνικό δημόσιο καλό εξ ονόματος όλης της κοινωνίας και να μην εκπροσωπούν απλώς τις κυβερνητικές αρχές. Συζήτησα τα ζητήματα αυτά με κάποιους επικεφαλείς εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και οι επαφές αυτές με ενθάρρυναν μπορώ να σας πω γιατί από τις 27 εθνικές στατιστικές υπηρεσίες ορισμένες έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο δύναμης, ευρωστίας, σεβασμού, ποιότητος. Δεν μπορούμε όμως να πούμε κάτι ανάλογο για όλες τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω στο προβλεπόμενο αυτό σύστημα, προκειμένου να έχουμε έναν μηχανισμό ο οποίος θα προβλέπει τους διευθυντές και διαχειριστές των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών. Ένα μηχανισμό ο οποίος θα πρέπει να ενδυναμωθεί και θα πρέπει ουσιαστικά ο άνθρωπος αυτός, επικεφαλής μιας στατιστικής υπηρεσίας, να έχει το ίδιο καθεστώς με αυτό το οποίο ισχύει για τον διοικητή μια κεντρική τράπεζας. Για ποιο λόγο θα πρέπει να προβλέπετε κάτι διαφορετικό. Και θα πρέπει να λογοδοτεί και στα κοινοβούλια και όχι μόνο στα Υπουργεία, ο επικεφαλής αυτός της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι πόροι των υπηρεσιών αυτών, προκειμένου πραγματικά οι στατιστικές υπηρεσίες να μπορούν να είναι αυτόνομες, να έχουν το δικό τους το προπολογισμό και να μπορούν να λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο ανεξάρτητα από τις εθνικές κυβερνήσεις. Και θα πρέπει επίσης να δούμε και ποιες διαδικασίες ακολουθούνται για την κατάρτιση των στατιστικών δεδομένων. Και πρέπει να δούμε επίσης και ποια είναι η μέθοδος η οποία ακολουθείται για την παραγωγή, την διάχυση, τη διαβίβαση των στατιστικών δεδομένων, ποιε είναι κατευθυντήρες γραμμές οι οποίες ακολουθούνται, ποια είναι τα πρότυπα. Καταρχάς πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με το επίπεδο το οποίο θέλουμε για τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και την ίδια τη Eurostat. Στα πλαίσια του συστήματος θα πρέπει να δυναμώσουμε και τους ε, κανόνες κατηγοριοποίησης ε, συγκεκριμένων ε, στατιστικών δεδομένων, τους ορισμούς που χρησιμοποιούμε, τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα στατιστικά δεδομένα και σε όλα αυτά τα ζητήματα της προστασίας των στατιστικών δεδομένων. Επαναλαμβάνω ότι δεν επικρίνω αυτή τη στιγμή όλες τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες Απλώς πιστεύω ότι υπάρχουν ορισμένες που μπορεί να έχουν φτάσει σε αυτά τα υψηλά πρότυπα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε όμως ότι το σύνολο των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών θα φτάσουν στο ίδιο επίπεδο και ότι θα τηρούν, θα πληρούν αυτά τα υψηλά πρότυπα. Γιατί ξέρετε ότι μία λυσίδα τελικά είναι όσο δυνατή, είναι και πιο αδύναμος της κρίκος. Και αν υπάρχει ένας αδύναμος κρίκος, αυτό επηρεάζει τελικά όλο, όλη την αλυσίδα, όλο το σύνολο του δικτύου. Πρέπει λοιπόν όλη η κρίκη της αλυσίδας αυτής του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος να είναι ισχυρή. Να αναφερθώ σε συγκεκριμένε προτάσεις που ήδη υπάρχουν στην έκθεση και τις ε, οποίες προτάσεις θα ήθελα αυτή τη στιγμή να ενισχύσω μέσω τροπολογιών. Αναφέρομαι στην ε, ανεξαρτησία της Eurostat και των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών. Και θα πρέπει να μας απασχολήσει και ο κώδικας διοντολογίας, στα πλαίσια του οποίου θα πρέπει να αναφερόμαστε και πάλι στην ε, ανεξαρτησία. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να ενισχύσουμε το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα με μια πιο δεσμευτική νομοθεσία. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για αναθεώρηση των συνθήκων. Δεν προβλέπεται στο άμεσο μέλλον, αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον θα πρέπει να μας απασχολήσει. Αν πραγματικά θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα ανάλογο του συστήματος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τότε θα πρέπει μια αναθεώρηση συνθήκης κάποια στιγμή στο μέλλον να λάβει χώρα. Θα ήθελα να προσθέσω και μια ακόμα πρόταση, αυτή που έχει να κάνει με τις ετήσιες εκθέσεις. Ξέρετε ότι οι κεντρικές τράπεζες έχουν μια αιτήσια έκθεση, έχουν υποχρέωση υποβολής ετήσιας έκθεσης. Θα θέλαμε κι εμείς, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, να προβλέπετε μια τέτοια έκθεση στα πλαίσια της οποίας θα εξετάζουμε στο διάστημα ενός έτους πού είχαμε τελικά τη μεγαλύτερη επιτυχία, ποια δεδομένα παρήχθησαν, ποιες γενικές διευθύνσεις συνέβαλαν στην παραγωγή των στατιστικών δεδομένων, πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε σε αυτές τις ετήσιες εκθέσεις. Εκθέσεις που βασικά θα μας ενημερώνουν για το πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό κάθε χρόνο. Υπάρχει επίσης μια γενικότερη συνένεση για το ότι το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα θα πρέπει να ενδυναμωθεί. Οι προτάσεις μας είναι σημαντικές και νομίζω ότι θα πρέπει να τις εφαρμόσουμε. Ωστόσο θα πρέπει να ανοίξει και μια συζήτηση για το πώς θα εξελιχθεί το σύστημα αυτό στο μέλλον, στα πλαίσια μιας νέας οικονομικής διακυβέρνησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά έχω να σας πω. Κύριος Γκοζές έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιγητά, θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη για την απουσία της κυρίας Κράτσα, η οποία είναι συνεισηγήτρια, ε, ε η οποία είναι σκιώδης για το θέμα αυτό. Δεν μου έχει δώσει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές. Όπως συνήθως λέω για θέματα στατιστικών, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σας και θα στηρίξουμε την πρόταση που θα υποβάλλετε για να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές στατιστικές. Και όπως το υπογραμμίσατε κι εσείς, πράγματι είναι πολύ σημαντικό οι υπηρεσίες, οι εργαζόμενοι σε αυτές να καταλήξουν σε αξιόπιστα ε, στοιχεία τα οποία να μην εξαρτώνται από τον πολιτικό παράγοντα διότι είναι πολύ ενοχλητική αυτή η τάση των πολιτικών να τροποποιούν τα στατιστικά στοιχεία αναλόγως με τις επιθυμίες τους χωρίς όμως ε, να ανταποκρίνεται αυτό στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Γκοζές. Φίλιπ, σειρά σου νομίζω. Μετρούσα κεφάλια. 25 νομίζω βρισκόμαστε εδώ στην κύρια αίθουσα και 40 και διερμηνείς. Ευχαριστούμε τους διερμηνείς, διότι δεν έφυγαν και μας ανέχονται. Ευχαριστώ και τη Eurostat που βρίσκεται εδώ και έχει υπομονή. Δεν θέλω να σας ε, ανησυχήσω. Εάν νομίζετε ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξη η προσπάθειά σας, βεβαίως και θα σας βοηθήσουμε και θα κάναμε με το παν για να βελτιωθεί και να πετύχετε τις φιλοδοξίες σας. Είναι πολύ καλή η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τίνουμε να στηρίξουμε τις τροπολογίες που έχετε υποβάλει. Τώρα, αν θέλετε να τις πάτε σε ένα ε, παραπάνω επίπεδο, σε ένα υψηλότερο επίπεδο, ναι, ε, και εμείς μπορούμε να υποβάλλουμε παρατηρήσεις. Συμφωνούμε με την ανεξαρτησία της Eurostat. Πράγματι θα πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία, αλλά ποτέ δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι εξορισμού οποιοδήποτε, οποιοδήποτε οργανισμός που απαρτίζεται από ανθρώπινα όντα είναι εξορισμού ε, ε, απαλλαγμένος από λάθη και υπάρχει πλήρης εγγύηση για τις καλές του επιδόσεις πάντοτε. Αυτό δεν ισχύει. Βεβαίως θα πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία, θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι, ισορροπία και αφού αναφερθήκατε και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θέλω να σας πω ότι δεν χαίρομαι καθόλου με την πλήρη ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Διακυβεύεται η δημοκρατία όταν ένα θεσμικό όργανο με τόσο σημαντικό ρόλο έχει ακριβώς αυτή τη θέση, όπου δηλαδή κανείς δεν το ελέγχει. Ποτέ. Και καθημερινά είμαστε μάρτυρες του πειρασμού ε, που ε, νιώθει αυτό το θεσμικό όργανο για να ε, αυξήσει τις εξουσίες του και σε άλλα χωράφια. Επομένως, ναι, η υπερβολική ανεξαρτησία των θεσμικών οργάνων και της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας ε, δεν θα πρέπει να περιορίζει το δημοκρατικό έλεγχο. οι εκλεγμένοι σε μια δημοκρατία θα πρέπει να μπορούν να ελέγχουν αν καθορίσουμε τι θέλουμε να μετρήσουμε, τότε αυτό καθορίζει και το αποτέλεσμα που θα πάρουμε από τις μετρήσεις. Εάν, για παράδειγμα, θέλει κανείς να μειώσει το ενεργειακό του αποτύπωμα ή, θέλει να μειώσει τις ανισότητες στο εισόδημα, τότε πρέπει να βάλει αυτά τα κριτήρια στη μέτρηση και μάλιστα να μετρώνται με αξιόπιστο τρόπο. Δηλαδή, σε πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να, κατα... να καθορίζεται τι είναι αυτό το οποίο συλλέγεται ως πληροφορία. Και μετά από πλευράς μεθοδολογίας θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ο τρόπος συλλογής των στοιχείων είναι αξιόπιστος και σωστός για να μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτά. Από εκεί και πέρα θα πρέπει οι πρακτικές που ακολουθούνται να είναι δημόσιες και αρκετά ευανάγνωστες για τον μέσο άνθρωπο. Χρειαζόμαστε δηλαδή περισσότερη δημοσιότητα και ε, Επίσης πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ελέγχει την ποιότητα των πρακτικών αυτών, να υπάρχει ένας ποιοτικός έλεγχος δηλαδή από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, αξιολόγηση από ομολόγους, βέλτιστες πρακτικές. Ενδεχομένως αυτά δεν πρέπει να μπουν σε αυτόν τον κανονισμό. Να έχουμε ένα μοντέλο από πάνω προς τα κάτω με τη Eurostat, μπορούμε να έχουμε και διμερή συνεργασία να μοιραζόμαστε τις βέλτιστες πρακτικές και να έχουμε συμφωνίες αδελφοποίησης μεταξύ κρατών μελών και υπηρεσιών. Αυτά όλα μπορούν να εξεταστούν. Τώρα, ως προς την τροπολογία υπαριθμών 5, τη δική σας. Εμείς θέλουμε να ενισχυθεί η προσβασιμότητα στα στοιχεία να σας πω ότι παρεπιπτόντως συγκέντρωνα στοιχεία για μια ομιλία που έπρεπε να κάνω και βρήκα στα στοιχεία ότι η Eurostat είναι καταπληκτική ως προς τα δημόσια στοιχεία. Τα βρίσκει μέσω της μηχανής, μηχανής αναζήτησης του Google. Αν όμως θέλει κανείς να βρει στοιχεία του ιδιωτικού τομέα στη Eurostat, καλή του τύχη. Εγώ δεν ε, μπόρεσα από το χρηματοπιστωτικό τομέα, το μη χρηματοπιστωτικό τομέα, για τα νοικοκυριά. Δεν ξέρω καν πού μπορώ να βρω αυτά τα στοιχεία ε, στη Eurostat. Ελπίζω να τα έχει η Eurostat, αλλά δεν είναι καθόλου προσβάσιμα ε, και ευκόλως εντοπίσιμα. Δηλαδή πολλά μένουν να γίνουν προς την προσβασιμότητα στα στοιχεία από πλευράς Eurostat για τον ιδιωτικό τομέα να μην έχουμε κανόνες χωρίς να έχουμε θεσμοθετήσει κυρώσεις. Αλλιώς δεν θα μπορούμε να του επιβάλλουμε, να του θέσουμε σε ισχύ και ενδεχομένως ε, θα πρέπει να κάνουμε πιο αυστηρό το καθεστώς των κυρώσεων. Τι άλλα έχω σημειώσει. Τονίζω την ανάγκη για την καλή ροή πληροφοριών μεταξύ της SSS ε, και της Eurostat. Δεν έχουμε ολοκληρώσει την ε, άποψή μας για τα θέματα αυτά. Και τέλος, ως προς την, ε, το θεμητό διορισμό, δηλαδή την νομιμότητα του επικεφαλής, ενδεχομένως να υπάρχει ένα κατόφλι στις ψήφους. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Ο κόσμος των κεντρικών τραπεζιτών είναι ανδοκρατούμενος. Ο κόσμος της στατιστικής υπηρεσίας έχει μεγαλύτερη ισορροπία από πλευράς εκπροσώπησης των δύο φύλων. Αν ναι, θα πρέπει αυτό να φανεί και στις ε, ηγετικές θέσεις. Αυτά είχα να πω, όχι ως επίκριση, αλλά ως συμβολή στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπασέσκου, θέλετε να μιλήσετε. Όχι. Παρακαλώ εσείς. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρότι λοιπόν δεν είμαι σκιώδης συγητής ε, της ε, ομάδας μου, της ECR, περνάμε καλά εδώ, μας αρέσει, γι' αυτό ήρθαμε. Παρότι λοιπόν δεν είμαι εισηγητής, θα μου επιτρέψετε να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις και ορισμένες εξ αυτών θα είναι γενικής φύσεως, αλλά σας παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή κύριε Πρόεδρε Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σας πω ότι έχω δύο ομάδες παρατηρήσεων. Η πρώτη ομάδα, και εδώ πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τη θέση σας, Δηλαδή εσείς μιλήσατε για την ανεξαρτησία του συστήματος, κάτι που εγώ το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, υπογραμμίσατε το συντονισμό με τις ε, εθνικές αρχές και αυτό θα καταστήσει το ευρωπαϊκό σύστημα πιο αξιόλογο. Το θέμα είναι κατά πόσον ε, όλα αυτά ε, είναι εφικτά. Βεβαίως ε, και ε, συμμεριζόμαστε τη θέση σας, αλλά τα δεδομένα πρέπει να είναι αξιόπιστα. Εσείς αναφερθήκατε επανειλημμένα στην ελληνική περίπτωση και το δικό μου το ερωτηματικό είναι κατά πόσον θα μπορούσε κανείς να αποφύγει αυτό το ελληνικό παράδειγμα. Κατόπιν, ε, έχω και άλλες παρατηρήσεις όπως σας είπα Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω κατά πόσον οι εθνικές αρχές μπορούν ή επιθυμούν να ανταλλάσσουν αξιόπιστα στοιχεία. Γιατί στοιχηματίζω ότι οι εθνικές στατιστικές ε, υπηρεσίες ε, κάνουν τα δικά τους ε, τα, δικά, τα δεδομένα πιο ε, ενδιαφέροντα, πιο, πιο βελτιω, περισσότερο βελτιωμένα. Και κάτι άλλο. Είναι εφικτό το να επιβάλλει κανείς μια κοινή μέθοδο, η οποία μέθοδος ε, να είναι ε, χρήσιμη για τα κράτη-μέλη. Και δεν θέλω βέβαια να υπερβάλλω ούτε να δαιμονοποιήσω την ελληνική περίπτωση. Όμως ε, αμφιβάλλω κατά πόσο θα μπορέσουμε να αποφύγουμε κάτι σαν την ε, ελληνική περίπτωση στο μέλλον. Σε γενικές γραμμές ε, πάντως, ε, συμφωνώ με αυτά που είπατε στην αρχή της ομιλίας σας. Και πάλι λοιπόν, ε, η κυρία Φώτ είναι η σκιώδη εισηγήτρια της ομάδας μας. Αυτά που είπα εγώ είναι έτσι γενικότερες παρατηρήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον επιθυμεί να λάβει το λόγο. Κύριε Μπαχάτα. Επίσης, ε, σας δω συγγνώμη κυρία Μπαχάτα. Ξέρω ότι πρέπει να φύγετε αμέσως μετά τη συνεδρίαση. Ε, γι' αυτό λοιπόν για άλλη μια φορά ε, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και επίσης και για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθυνθώ στην Επιτροπή. Εγώ θέλω να περιστώ μόνο σε τέσσερα σχόλια, τα οποία όμως είναι σημαντικά κατά την άποψή μας. Το πρώτο σχόλιο αφορά την ανάγκη ε, να αναθεωρηθεί η υπάρχουσα ε, νομολογία για τα στατιστικά δεδομένα. Αυτό είναι απαραίτητο για να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση της διαχείρισης ε, και να υπάρχει εξυγχρονισμός των στατιστικών δεδομένων. Επίσης έχουν υπογραμμιστεί τα απαραίτητα στοιχεία στην έκθεσή σας. Έχουν γίνει και τα σχετικά σχόλια και βλέπουμε να υπάρχουν τρία βασικά στοιχεία να ε, διασφαλιστεί η εθνική ανεξαρτησία των Εθνικών Στατιστικών Ινστιτούτων και της Eurostat, να ε, διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός ε, συντονισμός με τα Εθνικά Στατιστικά Ινστιτούτα και επίσης οι εθνικές κυβερνήσεις να γίνουν και αυτές συνυπεύθυνες έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία των δεδομένων. Αυτά είναι τα νέα εργαλεία που αφορούν τις ε, υποχρώσεις. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τη Eurostat. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει αναλάβει να ενισχύσει την εθνική διακυβέρνηση και έχει σαγάγει ε, νέα στοιχεία στην πρόσφατη απόφασή της για τη Eurostat. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ε, ως ε, εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά στατιστικά δεδομένα. Όσον αφορά την, τον εξυγχρονισμό, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να, υπάρχει, να διασφαλίζεται η πρόσβαση στα δεδομένα, γιατί αυτό είναι η προϋπόθεση για να μειωθεί περαιτέρω το βάρος. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαμορφώνει μια σωστά ισορροπημένη φιλοδοξία που είναι παγιωμένη στην συνθήκη. Κατά τη δική μας την άποψη, η πρόταση αυτή προχωράει όσο είναι δυνατόν και προσπαθεί να διαφυλάξει ε, την διοκτησία όλων αλλά και τη συνεργασία μέσα στο ισχύον ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω ότι η συζήτηση του Συμβουλίου έχει προχωρήσει αρκετά και σχεδόν όλες οι προτάσεις μας ε, δυστυχώς ε, προσκρούν σε αντίσταση στα κράτη-μέλη και υπάρχει μάλιστα και ο κίνδυνος ε, αποδυνάμωσης ορισμένων διατάξεων. Γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή ε, βασίζεται στην ε, υποστήριξη της Οικονομικής Επιτροπής, ως συνήθως θα έλεγα. Και το τελευταίο μου σχόλιο αφορά το επίπεδο φιλοδοξιών που συζητήθηκε από τον εισηγητή και τον ε, πρόεδρο. Πρέπει να σας πω ότι εμείς ανησυχούμε για κάποιες μη ρεαλιστικές προσδοκίες και για τον κίνδυνο υπερφόρτωσης των διαπραγματεύσεων με αιτήματα τα οποία απαιτούν ε, θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν την τρέχουσα οδηγία. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι συμμεριζόμεθα απόλυτα το όραμα που υπάρχει για ε, ένα αποτελεσματικό στατιστικό σύστημα το οποίο θα καλύπτει όλο και περισσότερο τις αυξανόμενες ανάγκες για στατιστικά, στατιστικές πληροφορίες και θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που θα είναι συνδεμένες με την ποιότητα της παρεχόμενης πληροφορίας. Κατά την άποψή μας βέβαια, για να γίνει αυτό, ε, πρέπει να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν και οι μεταρρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Εάν λοιπόν κατορθώσουμε να διαφυλάξουμε τις φιλοδοξίες ε, της πρώτης επιτροπής, που θα αναδιαμορφωθεί από τη δική σας Επιτροπή, αυτή θα είναι μια επιτυχία και πάνω σε αυτήν θα μπορούμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις μεταρρυθμίσεις μας αλλά και την ε, μακροπρόθεσμη ε, πολιτική ε, που θα εφαρμόσετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ για όλα αυτά τα σημαντικά που μας είπατε. Καταγράφουμε τις παρατηρήσεις σας. Δεν είναι πρόθεση της έκθεσης αυτής να πάμε πέρα από τα όσα προβλέπει η συνθήκη. Ωστόσο, όταν μιλάμε για ανεξαρτησία θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι θα πρέπει η ανεξαρτησία αυτή να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες μεθόδους, όπως για παράδειγμα μέθοδος πρόσληψης των επικεφαλής των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών. Ο Φιλίπ Λαμπέρ, ενδεχομένως να μην το είπε βέβαια αυτό ακριβώς έτσι, πάντως μας είπε ότι δεν υπάρχει απόλυτο σεβασμός προς τους οργανισμούς εκείνους οι οποίοι είναι απολύτως ανεξάρτητοι, χωρίς λογοδοσία. Σαφώς θα πρέπει να υπάρχει μια λογοδοσία προς εθνικές κυβερνήσεις, αλλά παράλληλα και προς τα, κυβων... κοινοβούλια. Αυτό αποτελεί μια ειδοποιώ διαφορά. Έχοντας ασχοληθεί όμως περισσότερο με τις στατιστικές και έχοντας εξετάσει όλη αυτή τη νομοθεσία την οποία έχουμε εκπονήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέσω διαφόρων νομοθετικών πακέτων όπως το 6-pack και το 2-pack και τον πίνακα βαθμολόγησης καταλαβαίνετε ότι τελικά μία χώρα εξαρτάται πάρα πολύ από συγκεκριμένα στατιστικά δεδομένα, από το έλλειμμα ή το χρέος για παράδειγμα. και να είμαστε τόσο απόλυτοι βασιζόμενοι σε ένα στατιστικό δεδομένο τελικά, συντοποιούμε ότι τα στατιστικά αυτά δεδομένα ενδεχομένω να μην έχουν εκπονηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ότι ενδεχομένω το αποτέλεσμα που έχουμε στα χέρια μα να μην είναι το καλύτερο δυνατό. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να δώσουμε υπερβολική διακριτική ευχέρεια για τα στατιστικά δεδομένα. Σαφώς καταλαβαίνω ότι θα πρέπει εγκαίρως να υποβάλλονται κάποια δεδομένα, αλλά πολλές φορές αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας είναι προσωρινά, πράγμα το οποίο σημαίνει τελικά ότι αυτά τα στατιστικά δεδομένα είναι υποκειμενικά. Επομένω, πρέπει κανείς να κάνει συγκεκριμένα κάποιες εκτιμήσεις στη συνέχεια βασιζόμενος σε προσωρινά δεδομένα ή απουσία δεδομένων. για συγκεκριμένα στατιστικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα αυτά τα οποία υπερβαίνουν, ή μάλλον που τα οποία δείχνουν ότι ε, το χρέος βρίσκεται πάνω, το, πάνω από το 3%, θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, γιατί αυτά τα στατιστικά δεδομένα οδηγούν στη συνέχεια σε επιβολή κυρώσεων. Όσοι λοιπόν είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση αυτό των στατιστικών δεδομένων θα πρέπει να χαίρουν πλήρους εμπιστοσύνης. Θα πρέπει να είναι πραγματική επικεφαλής αξιόπιστων υπηρεσιών. Οι περισσότερες είναι, πολλές είναι, αλλά πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε 27 αξιόπιστες εθνικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό γιατί τα στατιστικά δεδομένα τα οποία παράγουν οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικότατες συνέπειες συνέχεια για τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν αναφέρθηκα και στο ελληνικό παράδειγμα, γιατί ένα στατιστικό δεδομένο μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι μια χώρα έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με το έλλειμμά τη και όλε οι υπόλοιπε αποφάσει λαμβάνουν υπόψη βάση τη πληροφορία αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να έχουμε αξιόπιστε εθνικέ ε, στατιστικέ υπηρεσίε, καθώ επίση και ικανού ανθρώπου που να δουλεύουν για αυτέ. Αυτά είχα να σας πω. Κοιτάξουμε τώρα λίγο το χρονοδιάγραμμα. Σε 9 μέρες, σε 8 μέρες στις 14 Νοεμβρίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Η εξέταση τροπολογιών θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 17 Δεκεμβρίου κατά πάσα πιθανότητα. Και μάλλον η έκθεση αυτή θα πάει στην Ολομέλεια του Μαρτίου του 2013. Για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας, αυτή θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου και την 5η, 15η Νοεμβρίου. Στην ίδια εβδομάδα δηλαδή έχουμε δύο συνεδριάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Λύεται η συνεδρίαση.